Äh, Ξεκινάει η συνεδρίαση. Έχουμε πρώτα απ' όλα τις ε, ψηφοφορίες, ε, τις διάφορες εκθέσεις. Η πρώτη φορά την συνδεδεμένη τηλεόραση. Ο κύριος Καβαντά έχει ζητήσει το λόγο επί της διαδικασίας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ σύντομα για την ψηφοφορία του 89. Πώς ακριβώς θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Τη διάβασα στα γαλλικά και, και έτσι και αλλιώς την ερμηνεύω εγώ. Γι' αυτό παρακαλώ να την ψηφίσουμε σήμερα την τροπολογία αυτή και να την αφήσουμε για την Ολομέλεια και να βρούμε μια εκδοχή που θα ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλετε εσείς. Μίλησα με τη συνάδελφο και έτσι όπως είναι διατυπωμένη η τροπολογία δεν γίνεται κατανοητή από κανέναν. Μπορείτε, αν δεν μπορείτε να μας το πείτε, προτείνω να τα αναβάλουμε για την Ολομέλεια. Αν μας τη διαβάσεις μπορεί να προσπαθήσουν οι διερμηνείς να τη μεταφράσουν για να την καταλάβω. Λοιπόν, χθε με ενημέρωσαν διάφορε ευρωπαϊκέ οργανώσει του οπτικοακουστικού τομέα ότι η τροπολογία μου, υπερθμόν 89, ότι στην γαλλική εκδοχή του είχε εσφαλμένα μεταφερθεί στα γερμανικά και στα αγγλικά. Δηλαδή σήμαινε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο εγώ εννοούσα. Γι' αυτό θέλω να αποκαταστήσω τα πράγματα. Πιστεύω πως όλα αυτά οφείλονται σε μια ε, διατύπωση που είχα κάνει και στη σχετική ε, ε, ερμηνεία και μετάφραση. Και αυτό περιπλέκει λοιπόν τις συζητήσεις μας. Θα ήθελα λοιπόν ενώπιόν σας και ενώπιον των συναδελφών να σας μιλήσω για την τροπολογία αυτή και να την διατυπώσω με τη μορφή προφορική τροπολογία για να διευκρινίσω και να αποσαφηνίσω την θέση μου. Εδώ τι σημαίνει η τροπολογία αυτή στην αρχική της εκδοχή. Τονίζει πω είναι απαραίτητο ο δημόσιος τομέας να μην εξαρτάται μοναδικά από τις διαφημίσεις προκειμένου να διατηρήσει την ανεξαρτησία του και καλεί τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν τις προσπάθειες χρηματοδότησης του εν λόγω κλάδου. Αυτό ακριβώς σημαίνει η τροπολογία που έχω καταθέσει και ευχαριστώ που το σημειώσατε τελείως. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Jetzt habe verstanden. Danke den Τώρα κατάλαβα, ευχαριστώ τους διερμηνείς. Νομίζω μπορούμε να ψηφίσουμε. Τώρα που κατάλαβα λοιπόν, θα ψηφίσουμε αυτό το οποίο κατάλαβα. Εάν μπορεί να μου το γράψει και κάποιος από τους διερμηνείς, να το ψηφίσουμε. Όταν θα φτάσουμε στην ψηφοφορία, παρακαλώ Ήδη διερμηνείς να μου επαναλάβουν αυτό το οποίο είπε ο κύριος Καβαντά στα ωραία αυτά αγγλικά και γερμανικά για να μην καταλάβουμε κάτι λάθος. Γιατί εγώ έχω καταλάβει κάτι τελείως διαφορετικό. Εντάξει, περνάμε τώρα στην ψηφοφορία. Μετά, ναι, ωραία. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Προφορική 1 υπέρ. Κατά. Ξανά. Προφορική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. 61. Πέρασε. Δώδεκα. Υπέρ 16 κατά, η κυρία Παλιαδέλη επίσης. Κατά, απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Προφορική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 73. Πέρας. 19 υπέρ, 10 κατά. Δεκτή. Προφορική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 75 υπέρ κατά αποχές δεκτή 76 υπέρ κατά αποχές δεκτή 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 υπέρ κατά αποχές δεκτή 80-81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. Την 82. έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Με συγχωρείτε, αλλά δεν σηκώνετε τα χέρια αρκετά ψηλά. Λοιπόν, 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές δεκτή 85 υπέρ κατά αποχές δεκτή 86 υπέρ κατά αποχές δεκτή προφορική 487 υπέρ κατά αποχές δεκτή 88 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 89 υπέρ. Τι είναι αυτό. Α. Ξανατε, ξαναδιαβάστε την αγαπητή συνάδελφοι και παρακαλώ ακούστε προσεκτικά όλοι. Λόγω των σφαλμάτων που υπήρξαν στα, γαλλικά, στα αγγλικά και στα γερμανικά σε σχέση με το πρωτότυπο κείμενο αναφέρω. Υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο δημόσιος τομέας να μην εξαρτάται αποκλειστικά από διαφημίσεις ε, στην τηλεόραση, προκειμένου να διατηρήσει την ανεξαρτησία του και καλεί τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν τις προσπάθειες δημόσιας χρηματοδότησης του εν κλάδου. Ευχαριστώ. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 90 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 91 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 92 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 98 υπέρ, κατά αποχές να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 98. Πέρας. Απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαλτεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 8 με 12 δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 113 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 114 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 115 υπέρ. Κατά αποχές. Να θα βαλτεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ναι. Άμα δεν σηκώνετε τα χέρια δεν σας βλέπω. Συγγνώμη. Δεκτή λοιπόν. 116 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 117 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 118 υπέρ. Κατά αποχές να την με αρχιτή ψηφοφορία. Πέρας. 14 με 15 απορρίπτεται. 119 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά αποχές. Να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 130 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 131 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 132 υπέρ, κατά αποχές να την επαληθεύσουμε. Άρχεται ψηφοφορία. 132. Πέρας. Δεκτή. 133 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 134 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 143 υπέρ, κατά αποχές υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 144 υπέρ, κατά αποχές ε, δεκτή. 145 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 146 υπέρ. Κατά αποχές. Να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. 146. Πέρας. Δεκτή 18 εναντί 10. 147 υπέρ. Κατά αποχές. δεκτεί. 148 υπέρ. Κατά. αποχέ, Δεκτή. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 6 υπέρ. Κατά. αποχέ, Δεκτή. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. αποχέ, Δεκτή. 9 υπέρ κατά αποχές θα την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας 17 με 12 δικτή 10 υπέρ κατά αποχές θα την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία α καταπίπτει α μάλιστα με συγχωρείτε 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προφορική 5 υπέρ, ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 19 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας Δεκτή. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 43 υπέρ. Κατά αποχές να την επαληθεύσουμε. 43. Πέρας. Απορρίπτεται. 11-17. 44 υπέρ. Κατά αποχές να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. 44. Πέρας. 13 15. 45 υπέρ. Κατά. εποχέ. Πρέπει να τα επαληθεύσουμε. Έρχεται η ψηφοφορία. 45. Πέρα. 17 11 δεκτή. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 48 υπέρ κατά αποχές δεκτή 49 υπέρ κατά αποχές απορριφθείται 50 υπέρ κατά αποχές δεκτή 51 υπέρ κατά αποχές απορριφθείται 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή τελική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέρας 24 υπέρ 4 κατά μία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία κάμερεβέρτ. Περνάμε τώρα στην έκθεση του κυρίου Παπα-Νικολάου. Σκουρία, μάλιστα, με συγχωρείτε. Με πρώτη τροπολογία είναι του κυρίου Παπα-Νικολάου. Μάλιστα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Τροπολογία 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 14 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 78 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 88 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 80, 15, 15 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 16 και 90 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 17 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 99 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προφορική 100 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 101 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 102 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 103 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 105 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 106 υπέρ κατά αποχές δεκτή 107 υπέρ κατά αποχές δεκτή 108 υπέρ κατά αποχές δεκτή 110 με συγχωρείτε 110 δεν επηρεάζεται αγγλικά τι κάνουμε μου. 111 υπέρ κατά αποχές δεκτή 112 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 113 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 114 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 115 υπέρ, κατά αποχές δε, απορρίπτεται. 116 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 117 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 119 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 120 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 121 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 122 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 123 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 24 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 124 υπέρ κατά αποχές δεκτή 125 υπέρ κατά αποχές δεκτή 126 υπέρ κατά αποχές να το επαληθεύσουμε 126 Αρχή η ψηφοφορία πέρασε απορρίπτεται 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 128 υπέρ κατά αποχές δεκτή 129 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 131 υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 134 υπέρ κατά αποχές δεκτή 135 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή 138 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 30 υπέρ, κατά αποχές, δεκτή. 139 υπέρ, κατά αποχές, δεκτή. 31 υπέρ, κατά αποχές, δεκτή. 141 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 142 υπέρ, κατά αποχές, δεκτή. 33 υπέρ, κατά αποχές, δεκτή. 143 υπέρ κατά αποχές δεκτή 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή 145 υπέρ κατά αποχές δεκτή 146 υπέρ κατά αποχές δεκτή 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή 39 υπέρ κατά αποχές δεκτή 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή 43 υπέρ κατά αποχές δεκτή 150 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία 150 πέρας απορρίπτεται με μία ψήφο 151 υπέρ κατά αποχές δεκτή 152 υπέρ κατά αποχές δεκτή 45 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία 45 πέρας δεκτή 46 πέρα κατά αποχές δεκτή 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή 154 υπέρ κατά αποχές δεκτή 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. 156. Πέρας. Απορρίπτεται. 157 υπέρ. Κατά. εποχέ, Δεκτή. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 54 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 56 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχέ, δεκτή. 58 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 60 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή περνάμε στην 66 υπέρ κατά πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 74 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία 74 ναι ναι πέρας δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 75 υπέρ κατά αποχές Απορριφθείτε. 12 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 76 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Ψηφίζουμε στην τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. «29 υπέρ, καμία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια». Οπότε, τέλος. End of the vote. We on to Τελείωσαν οι ψηφοφορίες, περνάμε σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης. Ο Μάρκος Κουρία Πρέπει να ψηφίσουμε τι πράγμα. Πρέπει να συμφωνήσουμε για να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ποιος είναι υπέρ. Ναι, ναι, είναι σημαντικό. Λοιπόν, παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Αν συμφωνείτε να το συζητήσουμε με το Συμβούλιο. Πέρας. ένας υπέρ. Κανείς κατά. Ωραία. Ναι, ναι, είναι σημαντικό. Περνάμε σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης. Ε, εθελοντικές δραστηριότητες στην Ευρώπη. Ο κύριος Κουρία έχει το λόγο. Μικρόφωνο παρακαλώ. Okay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 αναφορικά με τη συνολική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Χρονιάς 2011 αναφορικά με τον εθελοντισμό λάβαμε την ανακοίνωση της ε, Κόμισιον και πάνω σε αυτήν ε, βασιζόμαστε για μια πρώτη ανάλυση. Αυτό το οποίο εντυπωσιάζει ευθύς εξ αρχής είναι πως ε, η Κομισιόν μας λέει και θεωρώ ότι αυτό έχει εξάλλου αποδειχθεί σε όλους όσοι παρακολούθησαν αυτήν την χρονιά, την ευρωπαϊκή χρονιά, πως είχε θετικές επιπτώσεις του εθελοντισμού τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Υπάρχουν μια σειρά αποδείκτες που το καταδεικνύουν αυτό. Το πρώτο σημείο της εκθέσεως ε, σχετικά με τη θέσπιση της χρονιάς για τον εθελοντισμό ενεκρίθη από το Κοινοβούλιο και προέβλεπε ε, μια ελάχιστη αναρμόνιση σε νομοθετικό πλαίσιο επί ενός ζητήματος το οποίο μέχρι τώρα ρυθμίζεται από εθνικού, εθνική νομοθεσία που διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους. Αυτό αναφίβολα ήταν ένα σημείο σημαντικό διότι υπήρξαν κάποια κρατημέλη τα οποία για πρώτη φορά υιοθέτησαν ένα νομοθετικό κείμενο για τον εθελοντισμό τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού. Στην αρχή λοιπόν αυτής της χρονιάς υπήρχαν μόνο 12 κράτη που διέθεταν ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο και κατά τη διάρκεια της χρονιάς προστάθηκαν Λιθουανία, Σλοβακία και Σλοβενία, η Βουλγαρία τα ενέκρινε την επόμενη χρονιά, δηλαδή το 2012, μόλον ότι έτυχε επεξεργασία στο 2011 και υπήρξαν και μια σειρά από άλλες χώρες όπως Πολωνία, Αυστρία, Πορτογαλία που είτε ανανέωσαν ε, τον νομοθεσία τους για τον εθελοντισμό είτε υιοθέτησαν μια στρατηγική επί του ζητήματος για να καταστήσουν τον εθελοντισμό ένα εργαλείο πιο δυναμικό στις κοινωνίες τους και σε ένα πλαίσιο πιο ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύει την επιτυχία. Αυτό ήταν και ένα από τα πρώτα ζητήματα που είχαμε θέσει ως στόχο στην εκθεσή μα. Υπήρξαν επίση κάποιες χώρες οι οποίες ενέκριναν το εγχειρίδιο αναφορικά με τον υπολογισμό του εθελοντισμού, με την μέτρηση αυτού. Θεωρήσαμε ότι αυτό ήταν ένα σημαντικό στοιχείο για να αποκτήσουμε ένα μέτρο, ένα δίκτυο, θέλετε, ενιαίο, αντικειμενικό, για το πώς ε, θα πρέπει να προσανατολιστούμε στο επίπεδο κρατών μελών σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τον εθελοντισμό και θα έχουν ε, κάποιους κοινούς δείκτες αντικειμενικούς. Πολλά κράτη-μέλη λοιπόν ενέκριναν αυτό το εγχειρίδιο κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Χρονιάς του Εθελοντισμού 2012 είτε αμέσως μετά το πέρας αυτού αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μας κάνει να υπογραμμίζουμε με ιδιαίτερη χαρά αλλά και με ικανοποίηση το αποτελέσματα αυτής της Ευρωπαϊκής Χρονιάς του Αθλητισμού για να μην μακρηγορήσω διότι θα πρέπει με αυτή την ευκαιρία να ακούσουμε και τις απόψεις των συναδέλφων βάσει των εμπειριών που απέκτησαν κατά διάρκεια αυτής της χρονιάς και στο πλαίσιο μια σειρά από δράσεων που ανήφθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπό λοιπόν αυτή τη ανακοίνωση, η Κομισιόν περιλαμβάνει και κάποια αριθμητικά στοιχεία για ορισμένε παρεμβάσει ε, που έγιναν κατά τη διάρκεια του έτου, και θα ήθελα τώρα να ασκήσω κάποια κριτική θα έλεγα πάνω στο ζήτημα αυτό. Π.χ. αναφέρει η Κομισιόν ότι οι επισκέπτες της ιστοσελίδες της ε, ε, Ευρωπαϊκής Χρονιάς Εθελισμού ήταν ε, λίγο παραπάνω από 366.000. Διερωτώ αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορούμε να το θεωρήσουμε ως θετικό ή όχι. Εγώ έκανα μια σύγκριση και μόνο η Εθνική Υπηρεσία Νέων στην Ιταλία ε, έχει, έτυχε 100.000 επισκέψεων στο, στο σελίδα της. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο λοιπόν αυτό το στοιχείο που σας αναφέρει η Κομισιόν είναι θετικό, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει. Πάντα ανεβάζεται διαδίκτυο, αναρτήθηκαν 420 βίντεο. Αυτό είναι θετικό στοιχείο ή όχι. Ελπίζαμε για κάτι παραπάνω. Όπως και το βίντεο κλιπ του Ευρωπαϊκού Έτους Θελισμού, πάντα η Κομισιόν λέει ότι το είδαν 26.000 ε, ε, φορές πρόσωπα. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα στοιχείο που εκφράζει κάτι το θετικό ή πόρο απέχει από το επιθυμητό. Ίσως θα πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά και να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα στα κράτη-μέλη στο πλαίσιο των εθελοντικών υπηρεσιών των πολιτών μας ότι όταν αναλαμβάνουν κάποια δράση θα πρέπει να τις ενημερώνουμε για να προωθούν μέσω το διαδικτύου έτσι ώστε να υπάρχουν πιο πολλές επισκέψεις και κάποια παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόστηκαν στα επιμέρους κράτη-μέλη. Σε αυτήν την περίπτωση λαμβάνω υπόψη ότι η σύνοψη είναι σίγουρα κάτι το απαραίτητο, δεν μπορούμε να καταγράψουμε όλα όσα έγιναν σε κάθε κράτος μέλος, αλλά το γεγονό ότι ε, μια σειρά από δραστηριότητες σε όλα τα κράτη-μέλη ε, μια κάποια σημασία και συμμετοχής ε, είναι κάτι που μαρτυράει για μια ακόμα φορά την επιτυχία αυτής της χρονιάς του εθελονισμού στα κράτη μας. Έχω άμεση γνώση του γεγονότος διότι παρακολούθησα κάποιες εξελίξεις, κάποιες ε, εκδηλώσεις στην χώρα μου, στην Ιταλία. Αυτά που αναφέρονται εδώ είναι κάπως περιοριστικά, αλλά είναι προφανές ότι έγινε μια δουλειά ιδιαίτερα συνοπτική για την παρουσίαση του εγγράφου αυτού. Έχουμε και κάποια παραδείγματα πρωτοβουλειών που έγιναν σε δραστηριότητες ε, εμβληματικές όπως δράσεις καινοτόμες. Γι' αυτό είναι ένα ενδιαφέρον σημείο. Ίσως θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και μερικές ακόμα, αλλά είναι ένα στοιχείο που μας ε, δείχνει πώς ε, έγινε ορατό αυτό το γεγονός από πλευράς του κοινού. Και καταλήγω λέγοντας ε, με μία ακόμα ερώτηση, την οποία θα ήθελα να θέσω και προς όλους τους συναδέλφους. Όταν συζητήσαμε για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελονισμού, τονίσαμε ότι δεν θα πρέπει να είναι μια χρονιά εορταστική, αλλά αυτή η πτυχή του εθελοντισμού που είχε γίνει ιδιαίτερα αισθητή και είχε ζητηθεί από μια σειρά οργανώσεων που είχαν έρθει εδώ στις Βρυξέλλες αλλά και στα κράτη-μέλη και με ζητούσαν ότι αυτή η εμπειρία, του ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εθελοντισμό να μην κλείσει και να μην πάψει με τον εορτασμό του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού. Και εμείς είχαμε κάνει κάποιες προτάσεις για να συνεχιστεί αυτή πρωτοβουλία, όχι εμπειρία, συγγνώμη, όχι μόνο τα, σε, στα ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών. Νομίζω ότι η Κομισιόν εδώ δεν μας ε, διαφωτίζει ιδιαίτερα, δεν προτείνει κάποια συνέχεια. Φαντάζομαι λοιπόν ότι πέρα από τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Χρονιάς Θεωρισμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει το θέμα, το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, διότι θα έχουμε αφηγηθεί όλα αυτά στην, στους στο ζήτημα του εθελοντισμού, θα τους έχουμε δώσει την στιγμή της ε, διασημότητας, να θέλετε, αλλά μετά θα υπάρξει μια οπισθοδρόμηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάποια βήματα προ τα εμπρό και να καταλάβουμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεχίσει να ασχολείται και να ενδιαφέρεται με αυτά τα θέματα. Στο σημείο αυτό να σταματήσω, διότι επιθυμώ να ακούσω τις εντυπώσεις ε, και των συναδέλφων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και με βάση αυτά που ήταν εδώ στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Νεβεντελόβα. Vážení kolegovia, ja som veľmi rada, že ako Marko správne povedal, tak práve moja krajina napríklad patrí medzi... Κοιτάξτε, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη γιατί η χώρα μου είναι ανάμεσα σε αυτές που πέρασαν νόμο για τον εθελοντισμό κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού. Δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως ακόμα, αλλά πάρα πολλά έχουν γίνει για να προωθηθεί ο εθελοντισμός. Ε, όπως είπε και ο Μάρκο, θεωρώ πως έχει σχηματιστεί μια συμμαχία εθελοντισμού και αμοιβαίας συνεργασίας και έτσι πρέπει να δοθεί περισσότερος χώρος για αυτές τις δραστηριότητες και να δημιουργηθεί μια δομή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι μια θετική εξέλιξη και πιστεύω και ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η τάση και στο εθνικό επίπεδο. Για μένα ο εθελοντισμός είναι κάτι το οποίο γίνεται για τους άλλους ανθρώπους χωρίς κάποια προσδοκία ανταμοιβή. Και βεβαίω. Υπάρχουν και εθνικές και ευρωπαϊκές ενώσεις που θα βοηθήσουν τους ε, τρόπους ε, από πλευράς ε, κοινωνικής ασφάλισης. Πρέπει να δημιουργηθούν και άλλοι μηχανισμοί ε, βοήθειας και επιπλέον ήταν έκπληξη, έκπληξη για εμένα το ότι τα κονδύλια που διατέθηκαν για τους εθελοντές φορολογούνται. Αυτό μου προξενεί έκπληξη. Γιατί η δουλειά η δουλειά αυτή γίνεται χωρίς καμία προσδοκία ανταμοιβή. Οπότε θεωρώ πως ε, δεν θα πρέπει να υπάρχει και φόρος. Πρέπει επίση να γίνονται κάποιε επιπλέον δραστηριότητες για να βοηθηθούν οι εθελοντέ Γιατί, όπως είπα, δεν αναγνωρίζεται αρκετά αυτή η δουλειά και πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα νομικό πλαίσιο για τις εθελοντικές δραστηριότητες για να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τον εθελοντισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. φίλους εθελοντές. Ε, έχω και έναν φίλο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα Κανάρια νησιά και βραβεύτηκε με το βραβείο Καρλομάγνου φέτος. Κάτι το οποίο ε, οφείλεται στο ότι δραστηριοποιήθηκε σε μια, δραστηρι... σε μια οργάνωση που λέγεται Ευρωπαϊκός Διάλογος και προσπαθεί να προωθήσει όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, ε, διάφορα παραδείγματα που πρέπει να μας εμπνέουν. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι ο Μάρκος Κούρια ήταν ε, υπεύθυνος για αυτή την έκθεση γιατί ε, ξέρει πάρα πολύ καλά το θέμα αυτό και επιπλέον για την αναγνώριση του εθελοντισμού πρέπει να αναγνωρίσουμε την εμπειρία που αποκτά ο κόσμος μέσω του εθελοντισμού. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει σε ένα επίπεδο το οποίο αναγνωρίζεται και στηρίζεται επαρκώς. Συμφωνώ και εγώ. Κυρία Βαζιά. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχικά να ευχαριστήσω τον κύριο Σκούρια, τον εισηγητή μας, διότι συμμερίζομαι την ανάλυση του. Θα είμαι όμως ε, κάπως πιο σκληρή αναφορικά με τον τύπο. Νομίζω πως η έκθεση Κομισιόν είναι τουλάχιστον απογοητευτικό. Ιδιαίτερα σε σχέση με τις φιλοδοξίες που είχαμε προσπαθήσει να θέσουμε σε αυτήν την χρονιά του εθελοντισμού. Θα ήθελα για μια ακόμα φορά να επαναλάβω πως στα γαλλικά ο όρος volunteer ε, μεταφράζεται με την λέξη μπένεβολα και όχι βολονταριά. Ε, αυτό είναι ένα καθαρά γλωσσικό ζήτημα. Νομίζω, δεν ξέρω τι θα πρέπει να γίνει προκειμένου να αποκατασταθεί ο όρος στην γαλλική. Το ζήτημα είναι ότι το μπένεβολα αφορά την δωρεάν δράση αλλά και την εθελοντική δράση ταυτόχρονα ενώ ο Ροσβόλων Τωριά δεν έχει αυτό νόημα. Κλείνω την παρέθεση εδώ. Νομίζω ότι είναι θετικό το γεγονός ότι διάφορα κράτη απέκτησαν νομικά μέσα τα οποία επιτρέπουν ένα, μια καλύτερη ανάπτυξη των ε, σε δραστηριοτήτων. Ελπίζω πως αυτό θα μας επιτρέψει να προοδεύσουμε για ένα ευρωπαϊκό καταστατικό περί οργανώσεων και ενώσεων για να επιτρέψουμε μια παγκόσμια αναγνώριση των ε, δικτύων που αναπτύσσονται στην Ευρώπη. Θεωρώ πως από πλευράς ε, του ε, εθελοντισμού. Αυτή τη χρονιά, ε, αυτό το έτος εθελοντισμού ήταν κάτι το πολύ θετικό. Κρίνω πως ε, εδώ δεν πάμε ιδιαίτερα μακριά στα συμπεράσματα ειδικά. Όταν βλέπω στο παράρτημα 2 αυτά που περιλαμβάνονται στα πρακτικά τα γαλλικά εντυπωσιάζομαι διότι δεν έχει κανένα νόημα ενώ στην Γαλλία υπήρξε μια ουσιαστική δραστηριότητα στον τομέα του εθελονισμού και χρησιμοποιήθηκε σωστά, αποτελεσματικά και προς το διατεύθυνση. Νομίζω, όπως συμβαίνει συχνά με αυτές τις ευρωπαϊκές χρονιές, εντάξει δεν ε, ε, ε, μάλλον ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε περαιτέρω με τον κύριο Σκούρια και φοβούμε, επειδή υπήρξε συγγύδρια για το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών, πως ο απολογισμός είναι πολύ πιο καταστροφικός από τη στην περίπτωση αυτή και οι δύο αυτές ε, ευρωπαϊκές χρονιές θα έπρεπε να είναι ε, καλύτερα διασυνδεδεμένες αλλά αντιθέτως από ό,τι εμείς επιθυμούμε η Κομισιόν αρνείται να δημιουργήσει σχέσεις και δεσμούς ανάμεσα στα διαφορετικά ε, ευρωπαϊκά έτη διότι θα μπορούσαμε να συνδέσουμε και την ευρωπαϊκή χρονιά ανεργού γύρανσης διότι εδώ Τώρα απέχουμε από κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά είμαι απόλυτα απογοητευμένη ε, ό,τι αφορά την έκθεση της Κομισιόν επί του ζητήματος ε, και θεωρώ πως θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους ε, παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών και την Συμμαχία για την Ευρωπαϊκή και το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού που συστάθηκε και προσπάθησε να πάρει τα πράγματα στα χέρια της για να δώσουμε μεγαλύτερη προβολή και μεγαλύτερη δυναμική στο ζήτημα σε σχέση με τα όσα πραγματικά συνέβησαν κατά τη διάρκεια αυτού του Ευρωπαϊκού Έτους. Ευχαριστώ Κριστίν Βέρζια. Είπες πράγματα με τα οποία συμφωνώ. Μπέκα. Äh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Μάρκο Σκουρία. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ματιά σε ένα τομέα που μας απασχολεί. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια παρατήρηση αυτή της ε, σύνδεσης των ε, θελοντικών ε, ετών. Εγώ ασχολούμαι με την πολιτική των ηλικιωμένων και υπάρχει βεβαίως και εκεί πέρα η σύνδεση με τον εθελοντισμό. Υπάρχει στο ευρωπαϊκό επίπεδο η λεγόμενη AIDS Platform και υπάρχει πραγματικά κάποια συνέργεια. Επίσης θεωρώ πως η αξιολόγηση της εργασίας της εθελοντικής πραγματικά είναι κάτι το πάρα πολύ καλό και έτσι θα αυξηθεί νομίζω και η σημασία που αποδίδεται σε αυτήν και θεωρώ πριν πω τα επικριτικά τα οποία θέλω να πω νομίζω πως αυτό ήδη αρκεί. Είναι πραγματικά μεγάλη αξία στην οποία αποδίδουμε όλα αυτό το οποίο δεν βλέπω είναι το εξή. Τουλάχιστον στην Αυστρία έχουμε 50% του πληθυσμού που ε, κάνει κάποια θελοντική δραστηριότητα. Κατά κύριο λόγο όμως είδαμε τις υφιστάμενες οργανώσεις να δραστηριοποιούνται. Την πρωτοβουλία, τους πολίτες κτλ. Και αυτό το οποίο ελπίζα και δεν το βλέπω στην έκθεση και θα ήθελα να υπάρχει κάπως περισσότερο και δεν ξέρω αν μπορεί να με στηρίξει η Κομισιόν μέσω μιας αξιολόγησης είναι η επίδραση σε αυτούς που δεν είναι ήδη εθελοντές. Ήλπιζα δηλαδή να υπάρξει μια περαιτέρω κινητοποίηση. Α, πάντων δεν τα βλέπω όλα αρνητικά. Εκεί όπου συμφωνώ απολύτως είναι πως ε, πράγματι το ευρωπαϊκό πλαίσιο αυτό είναι. Σωστό, καλό είναι να αναμένουμε αυτές τις πρωτοβουλίες. Εγώ θα αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα. Π.χ. Αυτό το οποίο ονομάζουμε ασφάλιση για αστική ευθύνη στις ε, εθελοντικές δραστηριότητες είναι κάτι το πάρα πολύ σπάνιο. Εκατοντάδες χιλιάδες ε, κάνουν εθελοντικές δραστηριότητες και αν βλάψουν ε, ανθρώπινη ζωή ή κάποια υλικά πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους. Αυτά είναι τεράστια τα ποσά αν πρόκειται π.χ. για ένα ατύχημα με ανθρώπους. Αλλά θα ήθελα παρόλα αυτά να πω πως βλέπω πάρα πολύ θετικά αυτή την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Έτους. Θεωρώ πως πράγματι πρέπει να κάνουμε αυτές τις εξολογήσεις με τρόπο σκληρό και πραγματικά να γίνει μια κριτική αξιολόγηση. Ευχαριστώ. Μπορείς. Ja tak Πράγματι η προσπάθεια γίνεται για την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Έτους ε, Εθελοντικής Εργασίας. Είχαμε πάρα πολλές συζητήσεις στο σύνολο της Ευρώπης γύρω από τον εθελοντισμό. Πρόκειται για μια προσπάθεια η οποία πράγματι αξίζει και είναι χρήσιμο να καταλήξουμε σε ορισμένα συμπεράσματα από τις εμπειρίες που συλλέξαμε από διάφορες χώρες και στην Πολογία έγιναν αρκετές συναντήσεις. Είχαμε σχεδόν 12.000 Πολωνούς οι οποίοι πήραν μέρος στην οργάνωση των μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων. Και αυτό λειτουργήσε και σαν θα έλεγα ε, μια επιπλέον προσπάθεια έτσι ώστε ο κόσμος να ασχοληθεί περισσότερο με τα θέματα του εθελοντισμού. Μιλάμε για κάτι θετικό δηλαδή και η επιδίωξή μας έχει σαν στόχο κάτι το ιδιαίτερα θετικό. Νομίζω ότι αντίστοιχε είναι και οι εμπειρίες από τις υπόλοιπες χώρες. Θα πρέπει καταρχάς να προσδώσουμε μια διεθνή διάσταση θα έλεγα σε όλες τις εθελοντικές οργανώσεις έτσι ώστε οι οργανώσεις αυτές σε εθνικό επίπεδο να αρχίσουν να μάθουν να συνεργάζονται με οργανώσεις εκτός της χώρας σε ευρωπαϊκό καταρχάς επίπεδο. Θα πρέπει επίσης να ζητήσουμε από τα διάφορα κράτη-μέλη έτσι ώστε και ένα τμήμα των ε, δραστηριοτήτων και των εργασιών σε επίπεδο ε, των δημοσίων λειτουργιών, όχι μόνο του ιδιωτικού τομέα, να καλύπτονται από τη συμμετοχή εθελοντών πολιτών. Η φροντίδα των ηλικιωμένων. Κάποια εύκολα πράγματα μπορούν να αντακαλύψουν φυσικά οι εθελοντές. Ε, και να μην ξεχνάμε ότι έχουμε εν λειτουργία μια ενιαία αγορά. Στο εσωτερικό αυτής της ενιαίας αγοράς έχουμε συζητήσει τα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος και το ίδιο θα μπορούσαμε να κάνουμε και για τις εθελοντικές οργανώσεις. Οι οργανώσεις των εθελοντών στο σύνολο της Ευρώπης μπορούν να συνεργάζονται, μπορούν να αναζητούν συμμάχους δηλαδή στις διάφορες χώρες πρόκειται για δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να είναι και διεθνούς χαρακτήρα, ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου λοιπόν θα πρέπει να τις εντάξουμε στην έκθεση. Βασικό λοιπόν είναι το να χαρακτηρίσουμε την προσπάθειά μας αυτή και με χαρακτηριστικά διεθνή έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε πρακτικές, να μάθουμε από αυτούς οι οποίοι μπορούν πιο αποτελεσματικά να μας δώσουν κάποιες ιδέες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Νομίζω ότι το ευρωπαϊκό αυτό έτος έδειξε κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Οι εθνικές ρυθμίσεις είναι θα έλεγα κάτι το ιδιαίτερα θετικό για την συνδυτοποίηση του Ευρωπαίου πολίτη και των οργανώσεων των εθελοντών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι που η επόμενη έκθεση είναι κάτι το οποίο θα, το ληφθεί, υπόψη από τον Μάρκο. Ε, μια λευκή βίβλος για την εθελοντική προσφορά. Είναι κάτι το οποίο έχει ζητηθεί ιδιαίτερα. Να καταλήξουμε δηλαδή σε ένα ευρωπαϊκό καθεστώς, σε έναν ευρωπαϊκό κανονισμό για την εθελοντική προσφορά εργασίας και σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο συλλογικό. Θα πρέπει να συγκρίνουμε τις τυπολογίες, θα πρέπει να συγκρίνουμε τις στατιστικές. Οι συγκρίσεις τις οποίες κάνουμε μέχρι τώρα τις κάνουμε δυστυχώς ανάμεσα σε δυσανάλογα διαφορετικές καταστάσεις. Εμείς δεν αναζητούμε την ομοιογενοποίηση, αναζητούμε όμως τη συγκρισιμότητα. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και αν οι ρυθμίσεις τις οποίες προτείνουμε σε διάφορες ε, ε, πολιτικές μας επηρεάζουν την εθελοντική εργασία. Πρέπει πριν από οτιδήποτε άλλο να θεωρηθεί η προσφορά των ε, εθελοντών σαν μια μορφή συγχρηματοδότησης, συμμετοχή στη χρηματοδότηση για να μπορεί κανείς να παίρνει μέρος σε διαγωνισμούς που προκυρήσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το θέμα δεν είναι λοιπόν να κάνουμε ένα απολογισμό απλά για το 12. Πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο έστω και σε επίπεδο soft soft-low, έτσι ώστε να μην μείνουμε στη διαπίστωση αλλά να προχωρήσουμε στην ικανοποίηση των ετοιμάτων που εκφράζουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με την εθελοντική εργασία και να διασφαλίσουμε και τη διεθνοποίησή της. Είναι απαραίτητο επίσης να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή εθελοντική εργασία, η οποία μέχρι σήμερα δυστυχώς έχει παραμείνει ιδιαίτερος περιθωριακή. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω όλα αυτά που υπόθηκαν. Στο πλαίσιο του προγράμματος ε, για τη διαβίου μάθηση συζητήσαμε αυτό ακριβώς το θέμα. Το θέμα δηλαδή του εθελοντισμού, της εθελοντικής εργασίας dieses auch als im Rahmen der Kofinanzierung von Jugendprojekten να γίνει δεκτό και στο πλαίσιο της ε, συγχρηματοδότησης ε. θεωρώ πως και η Κομισιόν είναι διαδεθειμένη να το δεχτεί. Κάτι άλλο θέλω να πω. Πέρσι τον Δεκέμβριο είχαμε εδώ πέρα πάρα πολλούς ε, Γερμανούς νέους που είχαν έρθει εδώ πέρα, εθελοντές, ε, εκατοντάδες και μίλησα μερικούς από αυτούς και πραγματικά με συγκίνησε. Με συγκίνησαν κάποια πράγματα από αυτά τα οποία μου είπαν. Ένας νεαρός μου είπε πως μετά από το ένα έτος που πέρασε, δεν θυμάμαι πλέον σε ποια χώρα, κάπου μακριά, γύρισα σπίτι μου και ήξερα πού βρισκόμουν, ήξερα τι μπορώ να κάνω και ήξερα τι ήθελα να σπουδάσω, έκανα κάτι τελείως διαφορετικό και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι υπάρχει αυτή η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. Οπότε οι νέοι άνθρωποι όταν δεν ξέρουν τι θέλουν να σπουδάσουν ή δεν σπουδάζουν έχουν τελειώσει το σχολείο και τα λοιπά, κάνουν κάτι ένα χρόνο όχι μόνο για τον εαυτό τους αλλά για την Ευρώπη. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και να υπενθυμίσω πως υπάρχει στη Γερμανία μια πρωτοβουλία που είχε υπογράψει και ο συνάδελφος ο κύριος ε, Κονβεντίτ. για το ότι ο κάθε ένας στη ζωή του πρέπει να έχει κάνει μία φορά κάτι εθελοντικά. Πολύ καλή πρωτοβουλία. Είχαμε πάρα πολλού σημαντικού στη Γερμανία που υπέγραψαν, στην Ευρώπη. Θεωρώ πως στην έκθεση αυτή δεν πρέπει να αναφέρουμε μόνο τον εθελοντισμό για τους νέους, αλλά για όλες τις ηλικίε. Και είναι σωστή η παρατήρηση ότι δεν υπάρχει αυτή η, η σύνδεση. Δηλαδή όταν δεν είναι κανείς πλέον 28 ετών που σταματάει αυτή η ναι. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Θελισμού μπορεί παρόλα αυτά να προσφέρει πάρα πολλά. Και έχουμε στη Γερμανία μια υπηρεσία προσφέρει τις υπηρεσίες ε, των πιο ηλικιωμένων, για μηχανικούς, για τέτοιους ανθρώπους που μετά πάνε ας πούμε στην Αφρική με αναπτυξιακές ομάδες κτλ. μετά τη σταδιοδρομία τους. Και προσφέρουν σε πάρα πολλούς τομείς. Και αγαπητέ Μάρκο, πραγματικά πρέπει εδώ πέρα σε κάθε ηλικία να μπορεί κανείς να προσφέρει εθελοντικά και να έχει την ευκαιρία. Και πράγματι πρέπει να υπάρχει, όπως είπατε, αυτή η ασφάλεια για αστική ευθύνη, γιατί οι άνθρωποι πάνε τόσο ή άλλως εθελοντικά, απλήρωτοι, ε, μην καταλήγουν να διατρέχουν και κίνδυνο ε, αν μπλέξουν σε ένα τύχημα. Μάρκο λοιπόν, ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ε, η Κομισιόν είναι εδώ πέρα, αλήθεια. Να, εκεί στο βάθο μάλιστα. Παρακαλώ. Ο κύριο Μακδόναλντ ε, πρέπει να είναι Α, ωραίος. Μάλιστα, μα φέρατε τίποτα. Α, περίμενα να κάνω καφεδάκι τουλάχιστον. Ήλπιζα. Έτσι. Όχι, όχι χάμπουργκερ. Δεν ανήκω στην οικογένεια που πήγε στι Ηνωμένε Πολιτείε και ίδρυσε την αυτοκρατορία των Χάμπουργκερ. Σα ευχαριστώ αγαπητά μέλη, ευχαριστώ Πρόεδρε, Σα ευχαριστώ για τα σχόλιά σα. Ήμουν υπεύθυνο τη Task Force στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαχείριση του προγράμματο. Με χαρά ακούω ότι με γενικού όρου θεωρείται ότι ήταν σχετικά θετική η κατάληξη. Αυτή ήταν η πρόθεσή μας. Δεν θέλαμε εμείς αυτό το ευρωπαϊκό έτος να περάσει απαρατήρητο. Κάναμε ό,τι προσπάθεια μπορούσαμε έτσι ώστε να υπάρξει μια θα έλεγα διαρκής παρακαταθήκη από την προσπάθεια αυτή. Είχαμε περιορισμούς βέβαια, κάποια πράγματα τα οποία θα ε, μπορούσαν να καταστήσουν τη ζωή των εθελοντών ευκολότερη είναι εθνικές αρμοδιότητες και προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τις εθνικές αρχές έτσι ώστε να πάρουν μέτρα που θα διευκολύνουν τη δράση των εθελοντών και τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται. Είμαστε ευτυχείς γιατί αρκετά κράτη-μέλη χρησιμοποίησαν το ευρωπαϊκό έτος σαν μια ευκαιρία να ξεκινήσουν νομοθετική δραστηριότητα προς την κατεύθυνση που προανέφερα. Ακούστηκε και κριτική, όλος περιέργος. για τις αδυναμίες του ευρωπαϊκού έτους για τον εθελοντισμό. Θα έλεγα σε επίπεδο διαδικτυακό Πράγματι η παρουσία μας θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα θέμα δημοσιονομικό πριν από οτιδήποτε άλλο. Είχαμε αρκετά χρήματα για το ευρωπαϊκό αυτό έτος σε σχέση με άλλα, αλλά αυτά τα 11 εκατομμύρια που αφιερώθηκαν στην προσπάθεια αυτή και στις προπαρασκευαστικές δράσεις για, για μια ήπειρο 550 εκατομμυρίων κατοίκων είναι ένα μικρό ποσό. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε πάντως και θα πρέπει να συζητήσουμε αν ε, όλες οι 20.000 επι, ε, ε, επισκέψεις ας πούμε στα βίντεό μας ήταν μια θετική παρουσία γιατί χρησιμοποιήσαμε ακριβώς αρκετό χρόνο για να αγοράσουμε χρόνο προβολής. Κάποια άλλα σχόλια τώρα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τίθεται το θέμα της ασφάλισης. Θα ήταν ε, πράγματι χρήσιμο αν κάποιες πρωτοβουλίες ε, νομοθετικές θα μπορούσαν να αναλυφθούν έτσι ώστε να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό επίπεδο κάλυψης των συγκεκριμένων ε, συνθήκων και προϋποθέσεων. Δεν είμαι σε θέση εδώ να αναλάβω κάποια υποχρέωση, αλλά θα λάβουμε υπόψη μας απλά τις απόψεις σας. Γενικά θα ήθελα να πω ότι και τα σχόλια τα οποία έγιναν για τις περιλήψεις των δραστηριοτήτων μας, επισκοπήσεις των δραστηριοτήτων μας, πράγματι θα μπορούσαμε να γράψουμε πολύ περισσότερα πράγματα, κάναμε όμως μια επιλογή Προσπαθήσαμε για το αν θα αφήσουμε εκτός κάποιες δραστηριότητες. Χαίρομαι πάντως που τα πράγματα πήγαν καλά και μπόρεσαμε να σας δώσουμε στο ένα άρωμα του τι υπήρξε και συνέβη τον προηγούμενο χρόνο. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω στην παρούσα φάση. Και θα επιστρέψω στην Επιτροπή με τα σχόλιά σας για τα οποία σας ευχαριστώ. Marco, do you Μάρκο, θες να πεις κάτι. Κοιτάξτε, θα λάβω υπόψη τις προτάσεις οι οποίες ακούστηκαν. θα ήθελα η έκθεσή μου να τη συμμερίζονται όλοι οι συνάδελφοι, να είναι μια έκθεση όλων των συναδέλφων, χωρίς περιορισμούς και να λάβουμε υπόψη μας τις ανάγκες αυτού του τόσο ενδιαφέροντος και σημαντικού κόσμου, του κόσμου της εθελοντικής προσφοράς. Λοιπόν αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας έτσι ώστε στο μέλλον να μην ξαναγίνουν οι ίδιες παρατηρήσεις. Δεν ξέρω πότε θα παρουσιαστεί η έκθεση. Πάντως ε, νομίζω ότι η προοπτική μας θα πρέπει να είναι αυτή που προανέφερα. Η έκθεσή σου θα συζητηθεί τον Ιούλιο. Γιατί? Α, γιατί πρέπει να μεταφραστεί. Και θα ψηφίσουμε τον Σεπτέμβρη. Εντάξει. Και θα κάνουμε αυτό το οποίο αφήσαμε το πρωί για τον ε, προϋπολογισμό το θέμα. As some of you probably already know, uh, we don't have a draft budget. Σας ξέρετε δεν υπάρχει σχέδιο προϋπολογισμού και αυτό βέβαια σκαθερεί όλη τη διαδικασία. Και δεν έχει κάποιο νόημα να συζητάμε προϋπολογισμό που δεν έχουμε δει. Έχουμε λοιπόν κάποια προβλήματα γιατί δεν ξέρουμε το πλαίσιο εντός του οποίου κινούμαστε. Έχουμε κάποια πιλωτικά έργα και μετά θα περάσουμε στις προπαρασκευαστικές δράσεις κτλ. Έχουμε πολλά στοιχεία του προπολογισμού που τρέχουν παράλληλα. Έχουμε τα πιλωτικά έργα που ανέφερα, έχουμε τις τροποποίησεις του γενικού προπολογισμού και γνωμοδότηση για τις προτεραιότητες της Επιτροπής μας και λόγω του ότι δεν υπάρχει σχέδιο προβλησμού, δεν ξέρουμε τα περιθώρια και το τι ισχύει για την Επιτροπή μας. Αλλά δεν αναμένουμε μεγάλες αλλαγές και περιθώρια λιγμών και πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη όταν κοιτάμε τα ποσά. Με βάση τις προπαρασκευαστικές δράσεις αυτές Έχουμε αρκετέ. Κάποια από αυτά τα έργα συνεχίζουν. Η γραμματεία σας έχει μοιράσει υποθέτω όλες τις προτάσεις. Φαντάζομαι πως ο κατάλογος τώρα θα πάει στη γραμματεία του προϋπολογισμού και μετά ο Επίτροπος θα αξιολογήσει τις άτυπες αυτές προτάσεις και θα ενημερώσει για να αποφασίσει ο κάθε βουλευτής εάν θέλει να υποβάλει προτάσεις ως τροπολογίες του προπολογισμού και σημειώστε πως πρέπει να καταρθούν όλα αυτά ως κανονικές τροπολογίες του προπολογισμού. Αλλιώς είμαι στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε τα προ... προπαρασκευαστικές δράσεις και τα πιλωτικά έργα και σύντομα θα έχουμε και μία ημερομηνία για την πρώτη συνεδρίαση και βεβαίως τότε θα έχω και περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτά από μένα ευχαριστώ. Äh, Μια σύντομη παρατήρηση τυπική φύση. Νομίζω πω οι προτάσει μου φτάσαν με κάποια καθυστέρηση και δεν έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο. Θα ήθελα αυτό το σφάλμα να διορθωθεί. Ευχαριστώ. Okay, we will do it. Huh? Wir können das aufnehmen. Εντάξει, θα το πράξουμε. Ωραία, ωραία, ναι. Είναι άτυπες οι προθεσμίες, οπότε εντάξει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Υπάρχει αυτό το έγγραφο. Τώρα θα το δει η Κομισιόν και θα μας πει τι μπορεί να γίνει. Τι δεν μπορεί να γίνει. Τι μπορεί να γίνει. και θα μας ενημερώνετε βεβαίως. Κάθε φορά φοβάμαι πως τα μέλη της Επιτροπής Προπολογισμού θεωρούν πως είναι η σημαντικότερη επιτροπή και δεν χρειάζεται να ασχολούνται μαζί μας. Αυτή είναι η συμπεριφορά τους. So, then, uh, last time we have decided... Την τελευταία φορά αποφασίσαμε να δώσουμε εντολή στον εισηγητή να αποκαταστήσει όλες τις γραμμές του προπολογισμού να κόψει κάτι να πει κάτι και γνωμοδότηση αναφέρει τις πολιτικές μας προτεραιότητες οπότε δεν θα ψηφίσουμε πρόκειται για άτυπη ενημέρωση δεν θα ψηφίσουμε τώρα θα ψηφίσουμε μετά έχουμε δώσει εξουσιοδότηση στον κύριο Λόκεγκάρτ και να μην τρέχουμε τώρα Αύγουστο ε, για να συνεδριάσουμε. Νομίζω προτιμάτε να κάνετε διακοπές. Και βλέποντας και κάνοντας. Αλλά και το σχέδιο προϋπολογισμού μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτηση για τις ιδέες σας για πιλωτικά έργα και προπαρασκευαστικές δράσεις, αν το θέλετε. Αλλά δεν νομίζω κανείς να τα έχει όλα αυτά. Το αρχίσω εγώ να λέω τα δικά μου και εσείς τα δικά σας δεν θα αλλάξει τίποτα. Περιμένουμε να τα δει η Κομισιόν και μετά. Εντάξει, ωραία. Ωραία. Έχει να... να πείτε κάτι άλλο. Είναι εδώ κανείς, όχι. Είχαμε και τη συνεδρίαση των συντονιστών. Θα τα υπόλοιπα θα δείξω email σας. Ε, Υπάρχει τίποτα άλλο στο διάφορα. Όχι, ευχαριστώ. Καλησπέρα. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ και τους